Ευρωπαϊκή Νομικών Υποθέσεων έλεγξε την εντολή των Μαριάντα Κατάινεν Μητροφάνοφ και πρότεινε να ανανεωθεί η εντολή τους από τις 28 Φεβρουαρίου, 5 μάλλον, Μαρτίου 2018. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Οι εντολές αυτές επιβεβαιώνονται.